Okay, Μπορούμε να προχωρήσουμε λοιπόν στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ουσιαστικά θα συνεχίσουμε την ε, ανταλλαγή απόψεων ε, με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο, τον κύριο Ντομπρόφσκης και τον κύριο Τζεντιλόνη. Ε, τους ευχαριστούμε που είναι διατεθειμένοι να παραμείνουν άλλη μία ώρα για να συζητήσουμε ε, το, τα προσχέδια προϋπολογισμού για τις... Ε, χώρες της Ευρωζώνης. Ε, δίνω το λόγο λοιπόν τώρα στους ε, επιτρόπους, το πολύ έξι λεπτά στον καθένα και κατόπιν θα έχουμε 45 λεπτά ερωτήσεις και απαντήσεις με πέντε λεπτά για κάθε ερώτηση και απάντηση. Κύριε Τομπρόφσκης, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Ε, συνεχίζουμε λοιπόν τη συζήτησή μας ε, μετά από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Τώρα θα επικεντρωθούμε στις ε, δημοσιονομικές αποφάσεις. Η προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε την ευθυνοπορεινή δεσμή μέτρων στις 20 Νοεμβρίου πέρσι που συμπεριλαμβάνει γνωμοδοτήσεις πάνω στα προσχέδια προϋπολογισμών των κρατών μελών της Ευρωζώνης, καθώς και αποφάσεις για διαδικασίες απόκλησης για την Ουγγαρία και τη Ρουμανία. Γενικά, οι απόψεις μας ε, για τις δημοσιονομικές πολιτικές των 19 ε, ε, χωρών, χωρών της Ευρωζώνης προωθούν τις καλές δημοσιονομικές πολιτικές και στηρίζουν τον συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών στην ζώνη του ευρώ. Όπως γνωρίζετε, το Eurogroup υποστήριξε και τις απόψεις μας τον προηγούμενο μήνα και χαίρομαι που μπορούμε σήμερα να συζητήσουμε τα θέματα αυτά μαζί σας σήμερα, διότι ε, έτσι γίνεται πιο δημοκρατική όλη η διαδικασία. Γενικά έχουμε κάποιες ε, καλές ειδήσει. Για πρώτη φορά με το 2002, κανένα κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν βρίσκεται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Ε, το συνολικό χρέος της Ευρωζώνης πέφτει, εννέα χώρες ε, έχουν ονομαστικά πλεονάσματα, ε, ενώ εννέα χώρες αναμένεται ή βρίσκονται πάνω από τους δημοσιονομικούς τους στόχους, τους μεσοπρόθεσμους στόχους. Αυτή η γενικά θετική εικόνα είναι το αποτέλεσμα καλών δημοσιονομικών πολιτικών σε κάποια κράτη-μέλη που φρόντισαν να επισκευάσουν τη στέγη όσο είχε ακόμα λιακάδα, όπως λέμε. Ε, πιο σημαντικό είναι όμως ότι αντικατοπτρίζει τις υποστηρικτικές οικονομικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες που ε, κυριάξαν τα τελευταία χρόνια. Φτάνω όμως τώρα και στα όχι τόσο καλά νέα. Καταρχάς, ε, πέρσι είδαμε ε, ε, εξασθένηση της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας οικονομίας. Στην Ευρώπη είχαμε επιβράδυνση των εξαγωγών και μείωση της παραγωγής. Και οι θετικές ε, δημοσιονομικές ε, ε, εξελίξεις κρύβουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε κράτη-μέλη. Πιστώσαμε ότι εννέα χώρες συμμορφώνονται με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, δύο χώρες συμμορφώνονται γενικά, ενώ οχτώ βρίσκονται σε κίνδυνο για μη συμμόρφωση. Ε, επίσης έχουμε χώρες όπου η μείωση του χρέους ε, δεν γίνεται αρκετά γρήγορα. Το Βέλγιο, η Ισπανία και η Γαλλία ε, έχουν πολύ υψηλούς λόγους χρέους και ΑΕΠ, σχεδόν 100%, ενώ το χρέος της Ιταλίας ξεπερνάει το 136% του ΑΕΠ. Οι τέσσερις αυτές χώρες δεν εκμεταλλεύτηκαν τους ευίουνους καιρούς για να συγκυρίσουν τα δημοσιονομικά τους και το ε, δεν ε, έχουν σχεδιάσει ουσιαστικά μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής. Αυτό είναι ανησυχητικό. Το γενικό μας μήνυμα είναι ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη δημοσιονομική τους εργαλειοθήκη για να προετοιμαστούν για πιο δύσκολους καιρούς που έρχονται. Ε, Πώ ε, ε, ακριβώς θα το κάνουν αυτό εξαρτάται από την κατάσταση τη κάθε χώρας. Ε, για τις χώρε με υψηλά επίπεδα χρέους, η καλύτερη προετοιμασία είναι να μειώσουν το χρέο, ενώ για τα κράτη-μέλη που έχουν δημοσιονομικό περιθώριο θα πρέπει να το εκμεταλλευτούν. Πέρσι το φθινόπωρο, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Πορτογαλία και η Ισπανία υπέβαλαν προσχέδια προϋπολογισμού που δεν προέβλεπαν καμία αλλαγή πολιτική. Στην ε, περίπτωση ε, της Πορτογαλίας ε, υποβλήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου επικαιροποιημένο προσχέδιο προϋπολογισμού, ενώ εκδώσαμε γνωμοδότηση στις 15 Ιανουαρίου, όπου καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η Πορτογαλία προβλέπεται ότι θα σημειώσει επαρκή πρόοδο για μείωση του χρέους. Επιπλέον προβλέπεται εξισορρόπηση του προπολογισμού το 2020. Ταυτόχρονα οι δημόσιε δαπάνε ξεπερνούν αυτό που ε, συνέστησε το Συμβούλιο. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι υπάρχει κίνδυνος μη συμμόρφωση ε, με το σύμφωνο. Επιπλέον, ε, πέρσι το φθινόπωρο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο πρότειναν υιοθέτησαν συστάσεις για την διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος για την Ουγγαρία και τη Ρουμανία. Επιπλέον η Ρουμανία φαίνεται ότι ε, ξεπερνάει το 3% του ε, ΑΕΠ ε, όπως προβλέπεται από την συνθήκη. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση. Πάντως γενικά η παρούσα κατάσταση δίνει μια καλή εικόνα της ανάγκης να εκμεταλλευόμαστε τους ευίωνους καιρούς για να δημιουργήσουμε δημοσιονομικά αποθέματα. Τα κράτη-μέλη που το έκαναν αυτά έχουν περιθώριο στη διάθεσή τους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να κάνουν επενδύσεις και να αντιμετωπίσουν ε, μελλοντικέ προκλήσεις. Άλλα κράτη-μέλη που δεν κατέβαλαν καμία προσπάθεια θα πρέπει να ε, ενεργήσουν πιο προσεκτικά και να ε, μειώσουν το, το χρέος τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Περιμένω να ακούσω τις απόψεις σας. Ευχαριστούμε. Ο κ. τώρα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Έχω κάποιες παρατηρήσεις. Θα έλεγα όσον αφορά τα θετικά. Συνολικά, ε, το κρατικό έλλειμμα συνολικά για την Ευρωζώνη θα παραμείνει κάτω από το 1% του ΕΠ το 2020. Όπως το ακούσατε, καμία χώρα δεν βρίσκεται στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και εννέα χώρες αναμένεται να πετύχουν τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς τους στόχους μέσα στο 2020. Επιπλέον, το κρατικό χρέος για την Ευρωζώνη θα συνεχίσει να πέφτει περίπου στο 85% του ΑΕΠ το 2020. Από την άλλη, η οικονομική δραστηριότητα επιβραδύθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια και όπως αναφέρεται στις προβλέψεις μας του φθινοπόρου δεν αναμένεται να ανακάμψει σύντομα. Θα ενημερώσουμε βέβαια τις προβλέψεις μας τον επόμενο μήνα και δεν αναμένουμε όμως μεγάλες αλλαγές όσον αφορά αυτή την προπτική. Επίσης έχουμε και εξωτερικούς κινδύνους από αυτού Υπάρχει η υπογραφή του πρώτου σταδίου της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, που όμως δεν φαίνεται να φτάνει για να αλλάξει συνολικά η εικόνα. Επιπλέον, η βελτιωμένη δημοσιονομική εικόνα κρύβει μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών μελών όσον αφορά το χρέος, όσον αφορά τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους και όσον αφορά τα δημοσιονομικά τους σχέδια και προγράμματα. Η το διαρθρωτικό πρωτογενές ισοζύγιο ε, θα παραμείνει με θετικό πρόσημο, όπως επίσης ε, και τα διαρθρωτικά ισοζύγια, κάτι το οποίο είναι θετικό βέβαια ε, στο σύνολο για την Ευρωζώνη. Τώρα οι χώρες, κάθε μία χωριστά, πετούν διαφοροποιημένη προσέγγιση, όπως είπα και πριν, όμως με συντονισμένο τρόπο. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το περιθώριο που έχει κάθε χώρα και να αποφύγουμε προκυκλικά δημοσιονομικά μέτρα. Οι χώρες της Ευρωζώνης συμφώνησαν όταν συζητήσαμε για αυτό το θέμα το Δεκέμβριο που μας πέρασε. Ας δούμε τώρα λιγάκι και τα σχέδια τα δημοσιονομικά της κάθε χώρας. Όπως είπα, υπάρχουν νέα χώρες που συμμορφώνονται με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Δύο από αυτές, η Γερμανία και οι κάτω χώρες, ε, ξεκινούν με τα πρώτα βήματα για μια περισσότερο επεκτατική και δυναμική δημοσιονομική πολιτική. Αυτό θα στηρίξει τη δικιά τους οικονομική ανάπτυξη, όπως επίσης και την ανάπτυξη ολόκληρης της Ευρωζώνης, αλλά και ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και καλούμε τις γερμανικές και ολλανδικές αρχές να προχωρήσουν σε επιπλέον δαπάνες για να στηρίξουν τις επενδύσεις. Τώρα, ε, ποιες χώρες κινδυνεύουν από μη συμμόρφωση. Όπως ε, τονίστηκε, Υπάρχουν κάποιες χώρες που εξακολουθούν να έχουν υψηλά επίπεδα χρέους και βιωσιμότητας. Κυρίως το Βέλγιο, η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία δεν συμμορφώνονται ούτε με τις συστηνόμενες προσαρμογές για τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους, αλλά ούτε και με τα κριτήρια μείωσης του χρέους. Δεν υπάρχει καμία πολιτική, ούτε σχέδιο, ούτε προγράμματα για το, την Ισπανία και το Βέλγιο. Τώρα για τις άλλες ε, χώρες, Σλοβενία, Σλοβακία, Φιλανδία και Πορτογαλία, που επίσης έχουν κινδύνους μη συμμόρφωσης, η Σλοβακία και η Φιλανδία ήδη κατέβασαν το χρέος τους κάτω από το 60% του έπαιρνε, η Πορτογαλία και η Σλοβανία μειώνουν το χρέος τους επίσης με κάποια ταχύτητα και έχουν φτάσει και στο κύριο έλλειμμά τους κάτω από το 3% του ΕΠΑ. Επιπλέον όμως, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς μας κανόνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτές οι τέσσερις χώρες κινδυνεύουν να αποκλίνουν από τις απαιτούμενες προσαρμογές για να πετύχουν τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς τους στόχους. Αυτό το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε το Eurogroup ε, μερικές φορές δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τις προσπάθειες που γίνονται από τις χώρες αυτές και τα αποτελέσματα ε, που δίνουν αυτές όσον αφορά ας πούμε την μείωση του χρέους. Οπότε συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις που θα αποτελέσουν και μια ευκαιρία για να συζητήσουμε πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα από το δημοσιονομικό πακέτο οι χώρες μέλη με υψηλά επίπεδα χρέους πρέπει να συνεχίσουν τις ε, ε, πολιτικές τους και εκείνες που έχουν δημοσιονομικό περιθώριο πρέπει να το χρησιμοποιήσουν για να αυξήσουν τις επενδύσεις. Με διαφορετική βέβαια προσέγγιση, αλλά να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και να ενισχύσουμε τον συντονισμό των δημοσιονομικών μας πολιτικών. Ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Πρόεδρος. Περνάμε τώρα στις ερωτήσεις. Δύο λεπτά. Καλωσορίζω και ε, τους κυρίους κυρίους πρόσκες και Τζεντιλόνι. Σχετικά με την ιεράρχηση του Green Deal και τη χρηματοδότησή της. Η πρώτη ερώτηση. Τι νομιο, δημοσιονομικός θα έλεγα βάρος μπορεί να προκαλέσει στα κράτη-μέλη. Υπάρχει κίνδυνος για τα κράτη-μέλη να πετύχουν τους στόχους τους οποίους έχουν. Και δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων όταν παρέμβει στα πλαίσια και του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης πιστεύετε ότι θα δοθούν περισσότερες δανειοδοτικές δυνατότητες σε χώρες οι οποίες έχουν μεγαλύτερες δημοσιονομικές δυσκολίες. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Το δεύτερο θέμα για τον κύριο Τζεντιλόνι. Αναφερθήκατε στην αναθεώρηση του 2-pack και του 6-pack, του διπλού και εξαπλού πακέτου. Αν και σε ένα ικανοποιητικό βαθμό βρίσκεται η εφαρμογή τους. Κάποιοι κανόνες πιο ξεκάθαροι, κάποιοι κανόνες πιο κατανοητοί, πιο διαφανείς, αλλά όχι ασθενέστεροι, όχι λιγότερο αυστηροί τι ρόλο μπορεί να παίξουν αυτά τα δύο πακέτα έτσι ώστε να διευκολυθούν οι επενδύσεις και στις πράσινες τεχνολογίες χωρίς ε, να διαταραχθεί η δημοσιονομική πειθαρχία. Για τον Green Deal αναφερθήκατε και στη Ρουμανία. Είπατε ότι θα έπρεπε να διευρύνουν τις δημοσιονομικές παρεμβάσεις σε εποχές οικονομικής ισχυρής ανάπτυξης η προηγούμενη κυβέρνηση είχε αναλάβει την υποχρέωση να αυξήσει ε, κατά 14% τις συντάξεις. Θεωρείτε ότι υπάρχει ανάγκη να αναβληθεί ένα τέτοιο μέτρο ή αντίστοιχα μέτρα. Υπάρχει κίνδυνος για την Ρουμανία να μην πετύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. yes. Τώρα για το θέμα της χρηματοδότησης του Green Deal. Για να χρηματοδοτηθεί αυτό το πρόγραμμα, το πράσινο, εν περιπτώσει, θα χρησιμοποιηθούν οι επενδυτικές δυνατότητες που υπάρχουν και θα πρέπει να κινητοποιηθεί όπως είπα τουλάχιστον ένα τρεις για τα επόμενα δέκα χρόνια. Στο εσωτερικό τώρα αυτού του προγράμματος θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός για να υποστηριχθούν οι περιοχές οι οποίες θίγονται περισσότερο από τη μετάβαση όπως οι περιοχές με ανθραχωρικία σαν παράδειγμα. Σχετικά τώρα με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, ε, προτείνεται να υπάρξει το λεγόμενο mainstreaming και στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού και στα πλαίσια του προγράμματος InvestEU και στις δυνατότητες που παρέχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό φυσικά θα απαιτήσει και α, α, εθνικές συγχρηματοδοτήσεις και επίσης θα πρέπει να βρεθούν και άλλοι τρόποι αντιμετώπισης των αναγκών μέσω και της λεγόμενης ρήτρα της επενδυτικής που, ασχολεί, που καλύπτει τέτοιου είδους περιπτώσεις. Τώρα, για τα κριτήρια διανομής ή κατανομής, αν θέλετε, των πιστώσεων, σε τομείς όπως ο άνθρακας, ο λιγνίτης, επιφανειακές, επιφανειακά κοιτάσματα, κοιτάσματα άνθρακα. Εδώ τίθεται ότι οι φτωχότερες περιοχές θα λάβουν περισσότερα από ότι οι περιοχές οι οποίες έχουν υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη. Τώρα για την δημοσιονομική κατάσταση στη Ρουμανία Πράγματι η Ρωμανία δεν έχει κάνει τα βήματα σχετικά με τις αποφάσεις του Συμβουλίου σε ορισμένους τομείς και φαίνεται ότι ξεπερνά ε, την σχέση ε, του υπερβολικού ελλείμματος και έχει ξεκινήσει μια διαδικασία ελέγχου. Ε, σε σχέση τώρα με τη δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να υπάρξει μια συνολική άποψη, μια συνολική εικόνα δεν μπορούμε να απομονώνουμε εμείς μονομένα στοιχεία. Θα ήθελα να δούμε στη Ρουμανία και το θέμα των εσόδων, γιατί ακριβώς ε, το φορολογικό βάρος είναι ένα από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Τζεντιλόνι έχει να κάνει κάποιο σύντομο σχόλιο. Είναι σαφές ότι η χρηματοδότηση του Green Deal είναι μία πρόκληση. Ακόμα και στη δική μας ανάλυση ε, το 1-3 δεν είναι το ακριβές βέβαια ποσό των επενδύσεων το οποίο χρειάζεται. Είναι ένα τμήμα των επενδύσεων που χρειάζονται. Η σύνθεση αυτής της προσπάθειας θα είναι μια σύνθεση η οποία θα έχει διαφορετικές καταβολές. Ε, τα, οι πιστώσεις ε, θα προέλθουν από τα ευρωπαϊκά ταμεία, από τις εθνικές χρηματοδοτήσεις, από τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες, οι οποίες θα παίξουν σημαντικό ρόλο και ε, η πραγματική πρόκληση είναι το πώς θα μπορέσουμε να διευκολύνουμε και τη δημόσια αλλά κυρίως την ιδιωτική χρηματοδότηση, τις ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτή τη συζήτηση πρέπει να την κάνουμε τον επόμενο μήνα. Όχι σε σχέση με τους κανόνες τους δημοσιονομικούς, αλλά και σε θέματα φορολογίας και σε θέματα κρατικών επιδοτήσεων. Είναι σαφές να δώσουμε στους επενδυτές ε, μία σαφή εικόνα. Δεύτερον, υπάρχει ο κίνδυνος διάχυσης ε, των μακροοικονομικών μας στόχων. Είναι επίσης σαφές ότι αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο να χάσουμε εδώ μια κάποια ευκαιρία. Όταν ο πρόεδρος λέει ότι το Green Deal είναι η νέα στρατηγική μας για την ανάπτυξη, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η δυσκολία εδώ είναι μια σαφέστατη δυσκολία. Θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στην χρηματοδότηση του Green Deal και να συνδέσουμε τις προσπάθειες και διεύρυνση των επενδύσεων προς τον Green Deal. Αυτό όχι για να ξεχάσουμε τους μακροοικονομικούς στόχους, αλλά για να προωθήσουμε την ανάπτυξη στην περιοχή του Euro. Ευχαριστώ πολύ. Φερνάντες, S&D. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω ισπανικά. Τρει ερωτήσει έχω. Η πρώτη μου έχει να κάνει με το πλαίσιο δημοσιονομικών ρυθμίσεων που έχουμε στη διάθεσή μας πέρα από το πακέτο των 2, των 6, το σύμφωνο σταθερότητας κλπ. έτσι κι αλλιώς δεν έχει ενσωματωθεί στο κοινοτικό κεκτημένο. Οπότε τις επόμενες εβδομάδες, μήνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για την αναθεώρηση όλου αυτού του πλαίσιου δημοσιονομικών ρυθμίσεων και θέλω να σας πω ότι η δικιά μου πολιτική ομάδα αναμένει να έχουμε κάτι παραπάνω από απλώ ένα προβληματισμό για την κατάσταση. Στην προηγούμενη θητεία είχαμε διάφορα white papers, διάφορα έγγραφα προβληματισμού και τα χαρακτηριστικά ε, του σημερινού πλαισίου έχει σαν αποτέλεσμα να περιμένουμε κάτι παραπάνω από γενικό προβληματισμό. Κατά τα άλλα, την προηγούμενη εβδομάδα ε, παρουσιάστηκε ο μηχανισμός αυτός δίκαιας μετάβασης. Πέρα από τον οργανισμό αυτό για τη δημιουργία του Ταμείου, που προφανώς προβλέπει μια αναθεώρηση των κρατικών ε, ε, ενισχύσεων προτείνεται ένας μηχανισμός που λέει ότι να παρουσιάσει νέα νομοθετική πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την γραμμή αυτή του προπολογισμού. Και αν αναθεωρήσουμε τις διατάξεις έτσι όπως προτείνει η Επιτροπή για τις κρατικές ενισχύσεις, ελπίζω η Επιτροπή να προτείνει και στον ε, κανονισμό μια διαφορετική δημοσιονομική αντιμετώπιση και να ξέρουμε κατά πόσο στην ε, μετάβαση αυτή θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε το κόσμο και να υπάρχει μια διαφοροποίηση ανάμεσα στις πλούσιες και τις άλλες ε, χώρες. Και έπειτα για το δεξίδιο του άνθρακα πότε. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ντομπρόφσκης. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας αυτές. Καταρχάς, όσον αφορά το δημοσιονομικό πλαίσιο, ε, το αγγίξαμε αυτό και στην προηγούμενη συζήτηση. Να επαναλάβω τα βασικά θέματα. Αυτή τη στιγμή αναθεωρούμε την, τις δέσμες σε 2 και 6 μέτρων αντίστοιχα. Και αξιολογούμε τους ισχύοντες κανόνες ενώ θα ξεκινήσουμε και τη δημόσια διαβούλευση για τις πιθανές προσαρμογές των κανόνων αυτών. Θα ήθελα να τονίσω ότι είναι σημαντικό να υπάρξει συνένεση σχετικά με το που θέλουμε να καταλήξει. Δηλαδή, εάν ε, αλλάξουμε τους δημοσιονομικούς κανόνες, να έχουμε μια καλύτερη κατάσταση από αυτή που έχουμε αυτή τη στιγμή, αντί να ε, ε, τελματώσουμε επί χρόνια σε μια διχαστική συζήτηση. Θα πρέπει λοιπόν να είναι σαφές πού θέλουμε να πάμε. η έκθεση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου πιστεύω ότι αποτελεί πολύ καλή βάση για τη συζήτηση. Όσον αφορά την ερώτηση για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, ε, όπως ήδη αναφέρθηκε, πράγματι, Μια πτυχή της προσέγγισης είναι η δυνατότητα για τις χώρες ε, με ε, χαμηλότερο επίπεδο να χρησιμοποιούν ε, μεγαλύτερο ποσοστό των ε, πόρων. Και δεν αναφερόμαστε μόνο σε οικονομικούς τομείς εντατικής χρήσης άνθρακα. Μας ενδιαφέρει γενικά η κατανομή του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης. Ευχαριστώ, Πάολο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ο στόχος της αναθεώρησης είναι όχι μόνο να, να συζητηθεί το πώς λειτουργούν οι κανόνες ε, των ε, δεσμών 2 ε, και 6 μέτρων αντίστοιχα, αλλά να διαπιστώσουμε και τι αλλαγές μπορούμε να επιφέρουμε. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για μας να ε, εξετάσουμε τις πιθανές αυτές αλλαγές κατά τη διάρκεια της συζητήσης. Θα πρέπει να εξετάσουμε τις διάφορες θέσεις ε, που υπάρχουν εντός του Κοινοβουλίου, μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ ενδιαφερόμενων ομάδων δεν μπορούμε να προτείνουμε μία ε, πρόταση από την κορυφή προς τα κάτω ε, αν θέλουμε να έχει ε, πρακτικά αποτελέσματα. Αν είναι να αλλάξουν, κάτι, να αλλάξουν οι κανόνες, αυτό θα πρέπει να γίνει με βάση μια κοινή συζήτηση. Η δεύτερη μου παρατήρηση έχει να κάνει με τον μηχανισμό, ε, το συνοριακό μηχανισμό προσαρμογής ε, όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Το ε, συνοριακό τέλος. Έχουμε ξεκινήσει μια μελέτη αντικτύπου και μετά από την μελέτη αντικτύπου θα ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση αφοσιωμένη ειδικά στους τομείς ε, που θα συμμετέχουν σε αυτόν τον μηχανισμό προσαρμογής. Ποιοι, ποιους τομείς λοιπόν θα καλύπτει αυτός ο μηχανισμός. Θα μπορούσαμε ίσως ένα χρόνο από τώρα, αρχές του επόμενου έτους, να έχουμε σχετική πρόταση. Είναι πολύπλοκο μέσο και θα πρέπει να το εξετάσουμε από νομικής πλευράς ε, και να εξετάσουμε και το περιεχόμενο είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Σας ευχαριστώ πολύ. Λαμβάνοντας υπόψη την πίεση χρόνου και ότι στις 6 θα αποχωρήσουν οι διερμηνείς, θα ήθελα να καλέσω τους συναδέλφους να περιορίσουν τις ερωτήσεις τους στο 1,5 λεπτό και να, δίνω και να να κάνω και ένα σήμα στους ε, ε, επιτρόπους ώστε να μείνουμε κάτω από τα ε, δύο λεπτά για τις απαντήσεις. Λουίς Καρικάνο. Ευχαριστώ πολύ. Έχω δύο ερωτήσεις ε, στα ισπανικά. Το έργο σας είναι σίγουρα περίπλοκο. Οι κανόνες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου προσπαθούν να πετύχουν διαφορετικούς στόχους, εξυγέννηση των δημοσιονομικών μας, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις ε, χώρες που πρέπει. Μερικές φορές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να χρειάζεται να δίνει περισσότερο περιθώριο σε μια χώρα από ότι σε μια άλλη. Αλλά τώρα κάποιες χώρες χάρη στις λεκίστικες υποσχέσεις που έκαναν προσπαθούν να πετύχουν στόχους όχι μόνο χωρίς μεταρρυθμίσεις αλλά κάνοντας και πίσω σε μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει όπως στην Ισπανία για παράδειγμα με μεγάλες μακροοικονομικές ε, ανισορροπίας, απασχόληση λοιπά, Η κυβέρνηση κάνει τα ανάποδα από αυτά ε, που πρέπει και τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, για παράδειγμα, να την παίρνει πίσω. Εσείς κάνατε μια αρκετά ανησυχητική διάγνωση για την Ισπανία, ότι δεν τηρεί τους δημοσιονομικούς στόχους. Ο κύριος Ντομπρόφσκης είπε ότι δεν κάνει αυτά που θα έπρεπε να κάνει. Ο κύριος Τζεντιλόνι είπε το 2020 θα είναι μια χαμένη χρονιά για ανισορροπίες κλπ. Εσείς δεσμεύεστε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα προσφέρει ευελιξία όσον αφορά το έλλειμμα και το χρέος σε χώρες οι οποίες για λαϊκίστικους λόγους εγκαταλείπουν τις μεταρρυθμίσεις στην οικονομία και μάλιστα σε χώρες οι οποίες αντιστρέφουν την κατάσταση και πάνε πίσω σε σχέση με μεταρρυθμίσεις που είχαν ήδη γίνει αποδεκτές στο παρελθόν. Απάντηση. Ο κύριος Τοπρόφσκης, όσον αφορά την ευελιξία ε, σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις. Έχουμε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, έχουμε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ρήτρα δηλαδή τέτοια, που ακριβώς λέει ότι οι χώρες που προχωρούν σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μπορούν να επωφεληθούν από κάποια ευελιξία. Και κάποιες χώρες χρησιμοποίησαν αυτή τη ρήτρα. Βέβαια, η ρήτρα αυτή για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις δεν υπάρχει για να αντιστρέφονται οι καταστάσεις και να παίρνουν πίσω οι χώρες τις μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη κάνει. Όχι. Εννοείται. Έπειτα, όσον αφορά τα δημοσιονομικά σχέδια της Ισπανίας. Πρόσφατα είχα συνάντηση με τον κύριο Καλβίνιο για να συζητήσουμε τον προπολογισμό του 2020 και πώς έχει προχωρήσει το έργο. Ε, το Υπουργείο με διαβεβαίωση ότι θα συνεχίσουν βάσει των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων. Οπότε μην καταλήγουμε πρόωρα σε συμπεράσματα. Ας περιμένουμε την νέα κυβέρνηση να παρουσιάσει τα δημοσιονομικά της σχέδια και βάσει αυτών θα προχωρήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αξιολόγησή της. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ζεντιλόνη για απάντηση παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ναι, θέλω να προσθέσω μόνο ότι το καλό νέο είναι ότι από ό,τι φαίνεται τώρα έχουμε στην Ισπανία μια κυβέρνηση που έχει δημοσιονομικές ε, αρμοδιότητες και άρα μπορεί να παρουσιάσει έναν προϋπολογισμό. Κάτι το οποίο είναι θετικό τόσο για την Ισπανία όσο και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις συναντήσεις μου με την Ισπανική κυβέρνηση μέχρι τώρα, δεν ήταν ακόμα ξεκάθαρο πότε θα έχουμε αυτό τον προπολογισμό. Είμαστε πεπισμένοι ότι θα έχουμε καλό διάλογο. Και φάνηκε και από τι συζητήσει με την Αντία Καλβίνιο ότι υπάρχει προσανατολισμός για συμμόρφωση με τους γενικούς μας κανόνες. Αλλά είναι μια συζήτηση που θα γίνει περισσότερο σε βάθος εφόσον έχουμε στα χέρια μας το σχέδιο, την πρόταση προϋπολογισμού της Ισπανίας. Ξέρετε ότι η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πλήρη συνεργασία και διάλογος για την εξέβρεση κοινών λύσεων. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Επόμενη ερώτηση για Γιακελούνιας από τους Πράσινους παρακαλώ. Σύντομα σε σχέση με αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως σχετικά με τις συζητήσεις που γίνονται για τις διαδικασίες μακροοικονομικών ανισορροπιών. Δεν ξέρουμε σε ποια φάση βρίσκονται και τι ε, δυνατότητες έχουμε να πάρουμε μέρος στη διαβούλευση και τι δείκτες χρησιμοποιούνται για τα μη δεδομένα ή μη καταγεγραμμένα μέχρι τώρα νομισματικά μέσα τα οποία έχουμε. Θα ήθελα να σχολιάσω επίσης ότι η διαδικασία αυτή αν γινόταν πριν από 15-20 χρόνια αυτό θα δημιουργούσε προβλήματα ανισορροπιών και ίσως τα ωφέλη να μην ήταν πάρα πολύ μεγάλα για ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα, για το δεύτερο, τη δημοσιονομική βιωσιμότητα μακροπρόθεσμα στα πλαίσια του νέου πολιετούς δημοσιονομικού Ξέρουμε ότι σε ορισμένου τομεί πολλά ταμεία θα μειωθούν κατά 20-25% και σε συσχετισμό και με τις δημοσιονο... δημογραφικές συγγνώμη, εξελίξεις αυτό θα δημιουργήσει τρομερά προβλήματα και κάποιες χώρες θα επηρεαστούν. Αναφέρομαι στη Λετωνία και στη Λιθουανία. Ο κύριος Ντομπρόφσκης έχει το λόγο. σχετικά με τις μακροοικονομικές, τη διαδικασία αυτή για τις μακροοικονομικές ανισότητες. Προσπαθούμε ακριβώς να λειτουργήσουμε με σωστό τρόπο στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας και δεν διαβλέπω σύντομα κάποια αμίζωνα θα έλεγα αλλαγή στα πλαίσια των ατυπικών νομισματικών παρεμβάσεων και μέτρων. οι χώρες θα πρέπει να, να συνεχίσουν τις προσπάθειες μείωσης του χρέους. και τα αποτελέσματα θα πρέπει να είναι, θα έλεγα, τα αναμενόμενα. Αναφερθήκατε επίσης και στο αν είχαμε ευρωπαϊκό εξάμεινο πριν από την κρίση, πριν από 15 χώρες και αυτό θα είχε εντοπίσει ήδη από τότε είναι αλήθεια δημοσιονομικές ε, ε, ανισορροπίες σε κάποιες χώρες και θα είχε επίσης προκαλέσει μια επιδείνωση της κρίσης. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια αυτό και αυτό που ακολούθησε, η κρίση που ακολούθησε το αποδεικνύει. Τώρα η τελευταία σας ερώτηση για το πολιετές το δημοσιονομικό ε, νομίζω ότι δεν είναι αντικείμενο συζήτηση σήμερα. Έχουμε και το πλαίσιο του Brexit. Δημιουργείται ένα κενό. Εμείς προτείνουμε μειώσεις χρηματοδότησης παραδοσιακών δραστηριοτήτων όπως και η γεωργία αν και ε, να φτάσουμε στο 1.11 του ΑΕΠ για να καλύψουμε κάποια από τα κενά αυτά. Τώρα, οι, δημοσιο... οι δημογραφικές τάσεις φυσικά και τις λαμβάνουμε υπόψη σε σχέση με την μακρόχρονη αηφορία των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Δεν μπορεί να είναι κάτι που αγνοούμε. <coughs> Δεν έχω κάτι να προσθέσω σε αυτά που είπε ο Μπάλτης. Νομίζω ότι η συζήτηση που κάναμε και αυτή και οι προηγούμενοι δείχνουν ότι θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο τη συζήτηση αυτή περισσότερο για την αναθεώρηση και των δικών μας κανόνων και σε επίπεδο διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι διαδικασία ακολουθήθηκε ε, πώς ε, δημιουργήθηκαν και έτσι θα μπορέσουμε να βρούμε τι πιθανές αλλαγές μπορούμε να κάνουμε. Είναι σαφές ότι κάτι το οποίο λειτουργεί σωστά, ας πούμε το έλλειμμα, πώς μειώθηκε τα τελευταία χρόνια, και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι τομείς στους οποίους είναι σαφές ότι έχουμε λιγότερες δυνατότητες να πετύχουμε ε, συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτό αποδεικνύει ότι η συζήτηση που θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα θα είναι πολύ χρήσιμη. Ρινάλντι, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τους Επιτρόπους. Θα αναφερθώ στο Σύμφωνο Σταθερότητας θα ήθελα να ζητήσω κάποιες διευκρινήσεις. Εμείς γνωρίζουμε ότι το άρθρο 16, το τελευταίο άρθρο δηλαδή, προβλέπει ότι μετά από πέντε χρόνια λειτουργίας, δηλαδή από το 1η Ιανουαρίου του 2013, θα ενσωματωθεί στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Το ερώτημα που θέτω είναι το εξής. Γνωρίζετε ότι το άρθρο 2 του Συμφώνου Σταθερότητας προβλέπει ότι τα συμβαλόμενα μέρη εφαρμόζουν την συνθήκη αυτή σύμφωνα πάντα με τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται στο βαθμό που είναι συμβατό με τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Το ίδιο Fiscal Compact λοιπόν στο σημείο 3 λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πρέπει ε, να συνεργάζεται με τις εθνικές διοικήσεις. Εδώ υπάρχουν κάποια θέματα. Οι δύο συνθήκες μας, το Μάστριχτ και η Λισαβόνα, λέγουν στο 104C αγγλικό και 126 τέως 124 ε, της ε, ε, Λισαβόνας ότι ισχύει το 3%. Ισχύει λοιπόν το σύμφωνο, η συμφωνία για την σταθερότητα και την ανάπτυξη, το σύμφωνο αυτό ή ισχύουν οι συνθήκες. Πρέπει να διευκρινιστεί. Ευχαριστώ κύριε Τομπρόσκης. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Καταρχάς, ε, σε σχέση τώρα με τη μεταφορά ε, του, ε, του, του Συμφώνου για την Ανάπτυξη στο, στην Ευρωπαϊκή, αν θέλετε, στις Ευρωπαϊκές Συνθήκες. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να μεταφέρουμε ακριβώς τις βασικές αρχές αυτού του συμφώνου στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος από το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο προτιμά να κρατήσει την κατάσταση αυτή ελεγχόμενη από το, από το διακυβερνητικό σκέλος. Σχετικά τώρα με τα θέματα των, της ισορροπίας των δημοσιονομικών κανόνων, το 3%. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν αντιφάσεις εδώ. Το Σύμφωνο Σταθερότητας αυτού προβλέπει ένα εξισορροπημένο προϋπολογισμό στα πλαίσια ενός οικονομικού κύκλου, εφόσον δεν ξεπερνάει το 3%. Αυτό είναι κάτι ε, το οποίο θα έλεγα εξηγεί την προληπτική δράση την οποία προσπαθούμε να εφαρμόσουμε και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και βοηθάει τα κράτη-μέλη να προσαρμόζουν τους στόχους τους ε, με τους στόχους τους μεσοπρόθεσμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατάσταση φυσικά διαφέρει από χώρα σε χώρα, όπου στις χώρες υπάρχουν ε, ας πούμε σε κάποιες χώρες υπάρχει υψηλό χρέος, τότε τα μέτρα θα πρέπει να συνοδεύονται από δημοσιονομικά μέτρα αλλά κυρίως και από διαφθορτικές αλλαγές ενώ σε άλλες χώρες ε, δεν υπάρχει διαφθορτικό έλλειμμα πάνω από το 1% του ΑΕΠ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τζεντιλόνι. Δεν έχω πολλά να προσθέσω σε αυτά τα οποία είπε ο Μπάλτης. Η δυναμική των σχέσεων ανάμεσα σε μια κοινωνική λογική και σε μια διακυβερνητική λογική φαίνεται μέσα από το ερώτημα της ένταξης του Συμφώνου Σταθερότητας στο δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτός είναι και ο λόγος για τους οποίους η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν υποστηρίχθηκε πλήρως και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το θέμα παραμένει λοιπόν ανοιχτό, όπως και άλλα θέματα, όπως και ε, το θέμα του Ταμείου της Παγκοσμιοποίησης που θα συζητηθεί στο μέλλον εκ νέου. Περνάμε στον επόμενο ομιλητή από τους συντηρητικούς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά το σύμφωνο σταθερότητας. Θα ήθελα να μάθω με ποιο τρόπο ο στόχος ο οποίος υπάρχει να γίνει πιο απλό και πιο γρήγορο το σύστημα, έτσι όπως προβλέπετε. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε αν οι τροποποιήσεις αυτές θα είναι διακανονιστικού τύπου ή αν θα έχουν σχέση με κάποιες ρυθμίσεις στο εσωτερικό όμως ενός διακανονιστικού πλαισίου το οποίο θα παραμείνει αμετακίνητο. Δεύτερον, η εφαρμογή τέτοιων μέτρων δεν θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη πιθανώς να πάρουν, ε, μέρος, να πάρουν μέτρα συγγνώμη, ε, στην προσπάθεια ελέγχου δημοσιονομικού. Ε, και μία συμπληρωματική ερώτηση σε σχέση ε, με αυτά τα οποία χαρακτηρίζουν το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Από τη μία οι μειώσει στον τομέα της συνοχής και στον τομέα της γεωργίας, όπως είπε μόλις τώρα άλλωστε και ο κ. Ντομπρόφσκης, θεωρούνται δεδομένες. Από την άλλη τα ταμεία για το Ταμείο Μετάβασης είναι κάτι το οποίο για αντικειμενικούς λόγους θα αδικήσει, θα έλεγα κάποιες χώρες εις βάρος κάποιων άλλων. Μήπως θα μπορούσαμε να δούμε τι περιθώρια υπάρχουν ε, για την χειροτέρευση της κατάστασης από τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν μετά από τις περικοπές στη Γεωργία εις βάρος ορισμένων χωρών, των Μπρόφσκης. Καταρχάς, όσον αφορά το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ε, πράγματι πολλά υπόθηκαν, αλλά σε επικεντρωθούμε στην πτυχή που θίξατε εσείς, ε, την απλοποίηση και πιο καλή αποτελεσματικότητα. Πράγματι βλέπουμε ότι υπάρχει περιθώριο απλοποίησης ε, του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και αυτός είναι ο λόγος που εξετάζουμε ε, σοβαρά τις εξετάσεις ε, του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Να ξεφύγουμε από κάποιους ε, δείκτες που μπορεί να είναι πολύ καλοί στη θεωρία, αλλά είναι πολύ δύσκολο να εξηγηθούν. Και εκ των υστέρων φαίνονται και αρκετά αβέβαιοι. Δηλαδή, αν δούμε ποιε ήταν οι αξιολογήσει όταν λάβαμε τι αποφάσει και πώ φαίνονται τα πράγματα διαφορετικά, είναι τελείω ε, εκ των υστέρων είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση. Ε, θέλουμε λοιπόν ε, έναν δείκτη για τις δαπάνες και να συνδέεται αυτό με το χρέος. Ε, Επίση, όσον αφορά το Ταμείο Δίκαιη Μετάβασης, στο πλαίσιο του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου, ε, έχουμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό ε, και έχει συμφωνηθεί ότι δεν θα πρέπει το Ταμείο Δικές Μετάβασης να συστηθεί εις βάρος άλλων πολιτικών 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν ε, επιπλέον πέρα από την ε, παρούσα πρόταση του πολίτου δημοσιονομικού σχεδίου. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τσεντιλόνη. Είναι δύσκολο στην αρχή της συζήτησης αυτής για την αναθεώρηση να πει κανείς το πώς θα ολοκληρωθεί η διαδικασία και πώς θα υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις νομοθετικές ή κάποιες προτάσεις διερμηνευτικές θα έλεγα, οι οποίες θα έχουν και αυτές τη σημασία τους. Αν ενθυμηθεί κανείς την ανακοίνωση του 2015 για την ευελιξία και για τα θέματα σχετικά με το Σύμφωνο για την Ανάπτυξη. Τελικά θα δει κανείς ε, μετά από λίγους μήνες συζήτησης και δημόσιας διαβούλευσης ε, το ποιο είναι το αποτέλεσμα. Ο κύριος Φίτο ρώτησε να μάθει, ζήτησε να μάθει αν υπάρχει μια κάποια καθυστέρηση. Στόχος μας είναι να ξεκινήσει η αναθεώρηση αυτή το ταχύτερο δυνατόν. Το κάνουμε αυτό δύο μήνες πριν από τη γέννηση της ε, ίδιας της Επιτροπής, ε, της νέας Επιτροπής και το μήνυμα το οποίο έκανε η πρόεδρος της Επιτροπής στα πλαίσια των προγραμματικών της δηλώσεων που έστειλε η πρόεδρος ε, προσκάλεσε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να χρησιμοποιήσει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία για την επιτυχία του Συμφώνου Ανάπτυξης και Σταθερότητας. Σχετικά τώρα με μια άνηση κατανομή των πόρων για τη μετάβαση, νομίζω ότι αυτός είναι ένας κίνδυνος ο οποίος πράγματι υπάρχει. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τον αποφύγουμε τον κίνδυνο αυτό. Και νομίζω ότι στα πλαίσια της συζήτησης που έχει ξεκινήσει υπάρχουν επιχειρήματα τα οποία μας οδηγούν στο να αποφύγουμε τους κινδύνους αυτούς. Ο κύριος Γκουσμάου από την Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι η κατάσταση στο εσωτερικό της Ευρωζώνης από τη μία έχει σαν στόχο τη μείωση των δημοσιονομικών ελλημάτων και τη μείωση του χρέους ταυτόχρονα. Για να το πετύχει αυτό η Ευρωζώνη εφαρμόστηκαν πολιτικές με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, διαφωνούσε πολλές φορές, γιατί τα μέτρα τα οποία ζητήθηκε να εφαρμοστούν ήταν πολλές φορές ε, πολύ πιο απαιτητικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτά τα οποία πρότεινε. Και η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα αντιμετώπιζε ας πούμε την Πορτογαλία ε, σαν μια χώρα η οποία παρουσιάζει κινδύνους σε σχέση με τη δημοσιονομική κατάσταση. Αυτό δεν είναι σωστό. Θα πρέπει οι διάφορες χώρες να είναι ισότιμες μεταξύ τους. Ε, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα χορήγησης εξαιρέσεων από τους δημοσιονομικούς κανόνες και όχι αυθαίρετες μερικές φορές ρυθμίσεις στον τομέα των μακροοικονομικών ανισοτήτων ιδιαίτερα για τις χώρες οι οποίες ε, παραβιάζουν ε, και το ε, όριο των τρεχόντων λογαριασμών. Ακριβώς η Γερμανία έχει ένα εμπορικό πλεόνασμα 2% από το 2010. Πολλές φορές έχει φτάσει και στο 6%. Οι Ολλανδοί έχουν αντίστοιχες επιδόσεις στο εμπορικό ισοζύγιο που έχει φτάσει και το 9%. Τι θα κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν παραβιάζονται οι κανόνες σχετικά με τα εμπορικά θα έλεγα πλεονάσματα. Ο κύριος Ντομπρόφσκης. Καταρχάς, όσον αφορά την δημοσιονομική απόδοση της Πορτογαλίας όταν παρουσιάσαμε τη φθινοπορεινή δέσμη μέτρων ε, του ε, Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με τον ε, κύριο Τζεντιλόνι, νομίζω ότι ήμασταν σαφείς. Κάναμε τη διάκριση ανάμεσα στα διάφορα κράτη-μέλη ανάλογα με την κατάστασή τους. Τονίσαμε τα κράτη-μέλη υψηλού χρέους που δεν εκμεταλλεύτηκαν τις καλές εποχές για να μειώσουν το χρέος. Η Πορτογαλία δεν ήταν από τα κράτη που αναφέραμε. Ε, αναγνωρίζουμε ότι μειώνεται το δημόσιο χρέος και το έλλειμμα του προπολογισμού. Μάλιστα προβλέπεται του χρόνου μικρό πλεόνασμα όσον αφορά τις ε, μακροοικονομικές ανισορροπίες ε, και ε, τα πλεονάσματα των, του ισολογισμού είναι ακριβώς ο λόγος που η Γερμανία και οι κάτω χώρες βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και γιατί εξετάζουμε πιο προσεκτικά την, τις δημοσιονομικές πολιτικές στις χώρες αυτές. Επανειλημμένα έχουμε ε, πει στις χώρες αυτές ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε ε, το δημοσιονομικό τους περιθώριο, να προωθήσουν ε, τις επενδύσεις. Και φέτος περιμένουμε να δούμε σημαντικές δέσμες μέτρων με, με κίνητρα, κάτι που βρίσκουμε ιδιαίτερα επίκαιρο στο πλαίσιο του παρόντος οικονομικού κύκλου. Ευχαριστώ πολύ κύριε τον Ο κύριος Τζεντιλόνι έχει το λόγο, αλλά πρώτα θα ανακοινώσω ότι σταματάει η διερμηνία. Θα συνεχίσουμε στα αγγλικά. Uh, yes, the... As far as Portugal is concerned, I think I, I've said also in my uh, introductory remarks uh, that also the opinion we adopted in a Eurogroup about Portugal shows that there is uh,